θα πρέπει να εφαρμοστούν σκληρότερα μέτρα. Σας ευχαριστώ, Επίτροπε. Πέρας της συζητήσεως. Και τώρα έχουμε την προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά αφορά τη μακροπρόθεσμη φροντίδα για τους ηλικιωμένους. Πρώτα απ' όλα θα δοθεί ο λόγος στην εισηγήτρια και στην συντάκτρια Λίν ε, για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ. Ο λόγος που υπέβαλα την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα στην ημερήσια διάταξη είναι για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε έναν αντιλογικό κώδικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη φροντίδα στου ηλικιωμένου. Δεν μιλάμε για νομοθεσία εδώ, αλλά για ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Επί μακρόν, η αντιμετώπιση των ηλικιωμένων υπήρξε ανεπαρκή σε πολλούς τομεί. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πρώτα απ' όλα τι στοιχεία έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την παροχή φροντίδα στου ηλικιωμένου στα κράτη-μέλη. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο όσον αφορά τη διάδοση των βελτίστων πρακτικών. Βασικό τομέα που απασχολεί είναι ε, η κα, κακομεταχείριση των ηλικιωμένων, συναισθηματική, οικονομική, φυσική. Ας πούμε μια γυναίκα 93 ετών που πήγε σε οίκο ευγυρίας για μια εβδομάδα και μόνο και να επιστρέψει και επιστρέφει αφιδατωμένη δεν τη βοήθησαν καθόλου καν να πιει κάτι. Αυτή δεν είναι μεμονωμένη υπόθεση. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις αφυδάτωσης κακής διατροφής. Θα ήταν καλό όμως να έχουμε στοιχεία συγκεκριμένα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται σε αφιδάτωση ή κακή διατροφή. Εξίσου ενησυχητικό είναι και η χρήση, η αποφυγή των μέτρων για αναβίωση κάποιων ηλικιωμένων. Περνάνε μια έντονη κρίση, να αποφασίσουν κατά πόσο θα πρέπει να ε, χρησιμοποιηθούν τα τεχνητή, τεχνητές μέθοδοι επιβίωσης ή όχι. Δεν μπορεί να αποφασίζει η νοσοκόμα και δεν πρέπει να πιέζονται οι συγγενείς να υπογράψουν ένα χαρτί σύμφωνα το οποίο θα αποσυνδεθεί από το μηχάνημα ε, ο ασθενής. Αυτές οι εντολές λοιπόν για την μη προσπάθεια επιβίωσης υποστήριξη του ασθενού. Αυτό μη εντολή να μην γίνουν προσπάθειε αναβίωση. Και το άρθρο 2 εξάλλου τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αναφέρει στο δικαίωμα στη ζωή. Τι γίνεται με αυτό. Χαίρομαι που η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία υιοθέτησε έναν ευρύ ορισμό ε, τη κακομεταχείριση των ηλικιωμένων. Θα πρέπει σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώση να καθορίσουμε το βαθμό τη κακομεταχείριση και θα ελπίζω να μας δώσει πράσινη βίβλο σχετική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ίδιος ο Επίτροπος αναφέρθηκε στο θέμα. Πάρα πολλά φάρμακα που χορηγούνται, αντιψυχωτικά φάρμακα και αυτά είναι, γίνεται κατάξη αυτών. Χρησιμοποιούνται προς όφελος του προσωπικού πολύ συχνά και όχι για ε, το άτομο το οποίο περιθάλπεται. Αντίθετα, ε, δεν τους δίνεται ιατρική περίθαλψη στους ηλικιωμένους λόγω ηλικίας και μόνο πολλές φορές. Άλλο ένα λόγο για τον οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο για απόφαση επί της οδηγίας ισότιμη αντιμετώπιση για να μην υπάρχει διάκριση όσον αφορά προ αγαθά και υπηρεσίε και εκεί συμπεριλαμβάνεται και η υγειονομική περίθαλψη. Κάθε κράτο μέσο πρέπει να κάνει περισσότερα πράγματα, τόσο ώστε οι ηλικιωμένοι να μπορούν να υποστηριχθούν στι κατοικίε του, αν αυτό επιθυμούν. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν ε, ποια είναι τα προσόντα εκείνων που περιθάλπουν ηλικιωμένου, θα πρέπει να υπάρχουν και μηχανισμοί κατάλληλοι εκπαίδευσή του. Πολλά κράτη-μέλη έχουν κάνει περικοπέ όσον αφορά τα ειδικά γυριατρικά φάρμακα. Θέλουμε να ξέρουμε αυτό τι συνέπειε είχε όσον αφορά του ηλικιωμένου. Να μην λησμονούμε ούτε και την υποστήριξη και αναγνώριση που χρειάζονται οι ανεπίσημοι περιθάλποντε. Πολύ συχνά αυτοί φροντίζουν με ελάχιστη βοήθεια του συγγενεί του καθημερινά όλη μέρα. Λοιπόν, όλο ο τομέα ε, αυτό έχει αγνοηθεί επί μακρόν τη μακροπρόθεσμη φροντίδα. Ελπίζω ότι το προφορικό ερώτημα και το ψήφισμα θα μα οδηγήσει στο να δίνουμε στο θέμα την σημασία που το αξίζει. Πολύ συχνά ένα ηλικιωμένο χρειάζεται μακροπρόθεσμη φροντίδα και είναι δύσκολο ηλικιωμένοι να εκφραστούν και να επασπιστούν δικαιώματά του. Θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε μαζί του, ώστε να εισακουστεί η φωνή του και να μην λησμονηθεί. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο Άντορ, σας παρακαλώ να σεβαστείτε πάρα πολύ το χρόνο που σας διατίθεται, διότι θα πρέπει να επιτρέψουμε και στους διερμηνείς να τελειώσουν τη δουλειά τους. Κύριε Επίτροπε, έχει το λόγο. Uh, Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, τις επόμενες δεκαετίες με την άτομα τα οποία ζουν όλο και σε μεγαλύτερη ηλικία σε όλες τις κοινωνίες θα πρέπει να βρούμε τους καλύτερους τρόπους για να ζήσουν. Αυτός είναι ο στόχος και είναι κάτι το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε και μακροπρόθεσμα για τους ηλικιωμένους. Το Νοέμβριο του 2009 ζήτησε το Συμβουλίο από την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράση για το 2011 για την πρόθεση της υγείας, της ποιότητας της ζωής και της ε, αξιοπρέπειας για όλους τους ηλικιωμένους. Χαίρομαι διότι η ε, επόμενες προεδρίες, η Ουγγρική και η Πολωνική θα προσπαθήσουν να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ήδη έχουν ληφθεί διάφορες πρωτοβουλίες από την Επιτροπή για την παροχή υπηρεσιών υγείας μακροπρόθεσμα ποιότητας και για να συζητήσει το θέμα αυτό περισσότερο σε όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο βασίζεται στον ανοιχτό τρόπο συντονισμού που θέλουμε να κάνουμε για θέματα ε, που αφορούν τους ηλικιωμένους και θα πρέπει από κοινωνική πλευρά να μπορέσουμε να επιλύσουμε το πρόβλημα και να δούμε πώς τις διάφορες αδυναμίες θα τις διορθώσουμε. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές και αυτό αποτελεί τους κυρίους στόχους μας. Η Επιτροπή μπορεί να είναι καταλήτης για τις αλλαγές και μπορεί να υποστηρίξει τις εθνικές προσπάθειες προετοιμάζεται από τις υπηρεσίες μας για τις ε, ε, μακροπρόθεσμη φροντίδια του τους ηλικιωμένους ε, το σχετικό έγγραφο και η ανακοίνωσή μας θα εκδοθεί το 2011. Χθε η Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση για τον ορισμό του 2012 το Ευρωπαϊκό Έτος για τους ενεργούς ηλικιωμένους. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλους ε, σε όλες τις χώρες ε, την, ε, τον στόχο αυτό, να έχουμε ενεργούς ηλικιωμένους. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε οτιδήποτε και να παρουσιάσουμε προτάσεις πραγματιστικές στη διάρκεια του 2012. Σωστά είπατε, για να μιλήσω πιο συγκεκριμένα, στις περισσότερες χώρες το βάρος έγκυται στην ίδια την οικογένεια για τους ηλικιωμένους. Σε όλες τις χώρες οι γυναίκες μάλλον είναι αυτές που φροντίζουν παρά οι άντρες τους ηλικιωμένους. Ε, ανεπίσημα και θα πρέπει βεβαίως να βοηθούνται ώστε να μην υπάρχουν κινδύνοι κοινωνικού αποκλεισμού κανέναν. Για να μπορέσει να διορθεί αυτή η κατάσταση, τα κράτη-μέλη μαζί με τη θεσμικά όργανα θα πρέπει να δούνε πώς θα μπορέσουν να ε, αξιολογήσουν ε, τις ε, δεξιότητες και τα προσόντα που πρέπει να έχει κανείς για να αναλάβει τέτοιου είδους διαρτραστηριότητες που σήμερα αναλαμβάνουν οι γυναίκες. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες από όλους. Χαιρετίζουμε τις ε, πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και από τις διάφορες σχετικές οργανώσεις. Η Επιτροπή δεν ε, θα συστήσει παρατηρητήριο για αυτό το θέμα, αλλά το να μάθουμε ε, όλοι για αυτό το active aging είναι κάτι που θα μας βοηθήσει όλους. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω και το πρόγραμμα που υπάρχει για την ε, παιδεία των ελληνίκων και να πω ότι και το έτος 2011 θεωρείται ως έτος θελοντισμού. Η κυρία Λίνα ανέφερε και την ηθική πλευρά αυτού του θέματος. Αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα και συμμερίζομαι απόλυτα την ηθική πτυχή αυτού του ερωτήματος που τέθηκε. Πολλές φορές όμως πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν θέματα όπως αυτό το οποίο είναι ε, θέμα ε, το οποίο χειρίζονται οι διάφορε χώρες μέλη και δεν μπορούμε εμείς και δεν έχουμε αρμοδιότητες για αυτό το θέμα. Βεβαίως μπορούμε να αναλάβουμε διάφορες πρωτοβουλίε όπως ένα συνέδριο που οργανώθηκε το Μάρτιο το 2008 το 2009 επίσης η Επιτροπή ε, εφάρμοσε ένα πιλωτικό πρόγραμμα που κατέληξε σε δύο project για να δούμε πώς μπορούμε στα διάφορα συστήματα υγείας να ε, κάνουμε κάτι καλό για τους ηλικιωμένους και του χρόνου των ε, φθινόπωρο θα παρουσιάσουμε και διάφορα πορίσματα μελετών. Επίση, μπορούμε στα πλαίσια του προγράμματο Δάφνη και στα προγράμματα δημοσία υγεία να χρηματοδοτήσουμε διάφορε εκθέσει. Υποστηρίζομαι τι εργασίε που γίνονται στα πλαίσια τη Επιτροπή Κοινωνική Προστασία για τις εθελοντικές κοινωνικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά ευέλικτοι ώστε τα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και στι διάφορες κοινωνικέ υπηρεσίες να παρέχονται εθελοντικά εκεί που θα μπορούσε να εφαρμογεί το ε, πλαίσιο προγράμματος θα είναι η μακροπρόθεσμη φροντίδα. Αυτό όμως δεν είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο και ξέρουμε ότι πολύ συχνά ε, τα άτομα τα οποία αφιερώνονται σε τέτοιου είδους ε, φροντίδες εξαιτία των υποχρεώσεων που έχουν πρέπει να εγκαταλείψουν όποια άλλη δουλειά θέλουν. Και βεβαίω εδώ τίθεται και θέμα εισοδήματος και συντάξεων αυτών των ατόμων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορεί κανεί ε, να συγκεράσει την επαγγελματική και την οικογενειακή του ζωή. Και ξέρουμε ότι πόσο δύσκολο είναι αυτό για τα άτομα που παρέχουν ε, άτυπα τέτοιου είδου φροντίδες στην οικογένειά τους. Θα πρέπει τα άτομα αυτά Επίσης να συμπεριληφθούν στα συστήματα κοινωνικής προστασίας πράγμα το οποίο θα ενθαρρύνει όλο και περισσότερα άτομα να προερέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Σε μία πρόσφατη μελέτη εξετάστηκαν όλα αυτά τα προβλήματα και είδαμε ότι Υπάρχουν διαφορές στα εισοδήματα και οι διαφορές σε επίπεδο φροντίδας είναι κάτι το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα δεδομένου ότι τα συστήματα διαφέρουν. Αυτό το οποίο ζητούμε είναι να γίνει περισσότερες έρευνες και πιο καινοτόμες πολιτικές στον τομέα αυτό και να προωθήσουμε σε όλες μας τις ε, πολιτικές μας, τις πολιτικές υγείας που είναι στρατηγική σημασία για τον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και τώρα οι διάφοροι εγωρητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Σόγκορ ε, για δύο λεπτά, μέσα του ΕΛΚ. Η γύρανση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μεγάλο πρόβλημα σε όλα τα κράτη-μέλη. Και πρέπει να τονίσουμε περισσότερο τη βελτίωση της φροντίδας για τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις φροντίδας ηλικιωμένων στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες όπου πολλές ε, γενναίες συμβιώνουν και λύνουν μέσα στο ίδιο νοικοκυριό πολλά από αυτά τα προβλήματα. Στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες ε, η φροντίδα είναι, σε, είναι πιο ιδρυματοποιημένη. Η, στο φως της οικονομικής κρίσης ε, η φροντίδα στα ιδρύματα αντιμετωπίζει προβλήματα και λόγω της γύρανσης του πληθυσμού. Στη χώρα μου οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι εκκλησίες και άλλοι οργανισμοί προσφέρουν φροντίδα αλλά πολλές φορές δεν τα καταφέρνουν και δεν υποστηρίζονται από την κυβέρνηση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έγινε πολλή δουλειά για να ε, απασχοληθούν αλλοδαπές γυναίκες μετά από επιμόρφωση στον τομέα αυτό. Είναι χρήσιμο αυτό το παράδειγμα από το οποίο μπορούν να διδαχθούν και άλλες χώρες. Εκτιμώ ιδιαίτερα την ε, το ε, αίτημα της Ελίζα Μπεθλίν. Η Κομισιόν θα πρέπει να καταρτήσει πράσινη βίβλο των πρακτικών για να διαλέγουν τα κράτη-μέλη τις καλύτερες, τις πιο αρμόζουσες στη δική τους πραγματικότητα, ούτως ώστε να, αποφεύγονται οι να αποφεύγεται η κακομεταχείριση δικαιωμένων. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές. Γκόντς για 90 δευτερόλεπτα. Κυρία Γκόντς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η αυξανόμενη μακροζωία είναι ένα επίτευγμα. Μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Ζουν περισσότερο οι άνθρωποι. Όμως είναι και πρόκληση. Πρόκληση διότι θα πρέπει να φροντίσουμε τους ηλικιωμένους σε μια γυράσκουσα κοινωνία. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την κοινωνική συμμετοχή των ηλικιωμένων. Να αποφύγουμε τη διάκριση κατά αυτών. Να αυξήσουμε τα χρόνια που ζουν υγιείς. Σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους δώσουμε συντάξεις. Το έτος ενεργού γύρανσης, active aging, μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση. Θα έρθει όμως η στιγμή όπου οι ηλικιωμένοι δεν θα μπορούν πλέον να φροντίσουν τους εαυτούς τους. Και αυτό αυξάνει τις δικές μας ευθύνες που πρέπει να τους παράσχουμε κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίδα κυρίως σε εκείνους που ζουν με χαμηλό εισόδημα. Μιλάμε για μέρημνα στο σπίτι ή σε κάποια ιδρύματα. Ζητούμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας βοηθήσει να τα πετύχουμε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα χρειαζόμαστε στοιχεία. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στις πλέον ευάλωτες ομάδες και να συλλέξουμε τις βέλτιστες προδιαγραφές για να καθορίσουμε τις ελάχιστες προδιαγραφές. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Η κυρία Λάμπερτ έχει το λόγο για ένα δίλεπτο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Λις Λίν για τη δυνατότητα που μας δίνει να συζητήσουμε το θέμα και καλωσορίζω πολλά από αυτά που είπε ο Επίτροπος. Αρκετά ενθαρρυντικά ήταν αυτά που είπε. Θα καταλαβαίνετε ότι κάποια θέματα που θυγούμε αφορούν τον ευάλωτο, το ευάλωτον κάποιων ηλικιωμένων και ότι θεωρούμε ότι είναι κρίσιμη σημασία να αισθάνονται ασφαλείς έναντι των των των ηλικιωμένοι. Βέβαια, εδώ πετύχθηκε το θέμα την αρμοδιότητα του κράτου μέλου. Η, η μέθοδο του ανοιχτού ε, συντονισμού υπάρχει, ούτω ώστε να μπορέσουν να εργάζονται τα κράτη-μέλη επί ενό θέματο που ναι, δεν είναι αρμοδιότη τη Ευρωπαϊκή Ενώση, αλλά θεωρείται κάτι που είναι από κοινού σημαντικό. Βασική φροντίδα, διατροφή, βασικά θέματα είναι και αυτά εντό αυτού του πλαισίου. Τι άλλα βήματα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πει στα κράτη-μέλη για το πόσο αποτελεσματική από πλευρά κόστου είναι η υποστήριξη των άτυπων περιθαλπώντων. Στο Ενωμένο Βασίλειο πιστεύετε ότι εξοικονομούνται δισεκατομμύρια από την οικονομία μας διότι η φροντίδα παρέχεται από φίλους, από συγγενείς και όχι από το κράτος. Και ότι η επένδυση σε κάποιο επίδομα εκείνων που φροντίζουν ή υποστήριξη σε εκείνων που φροντίζουν αυτό είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να γίνει. Αντί να απομονώνονται αυτοί οι άνθρωποι ε, και να υποφέρουν από μόνοι τους και να έχουν προβλήματα. Μάλιστα, περιθάλπουν άλλου και έχουν προβλήματα που δημιουργούνται του ίδιου γιατί έχουν κουραστεί και δεν τη χάνουν υποστήριξη. Και ποια δυνατότητα να βελτιωθούν τα προσόντα εκείνων που παρέχουν την υποστήριξη. Δεν είναι μόνο γυναίκες, πολύ συχνά είναι γυναίκες μετανάστες που παρέχουν αυτή την περίθαλψη και χρειάζεται επένδυση. Το ψήφισμά μας αναφέρεται και στην ανάγκη συμβάσεων που θα προβλέπουν ένα ελάχιστο ημερομίσθιο, ελάχιστη, ελάχιστο εισόδημα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Περιμένω σχόλιά σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, για τους μη εγγεγραμμένους. Στο Γιάννοφ έχει το λόγο για ένα λεπτό. κύριο στο Γιάννοφ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η... Τη γιαγιά μου τη γνωρίζω καλά. Ξέρω ότι οι ηλικιωμένοι θέλουν να φροντίζουν τον εαυτό τους όσο μπορούν. Όμως ο στόχος είναι ανέφικτος για πολλούς από αυτούς. Η μέση σύνταξη στη Βουλγαρία είναι 100 ευρώ. 100 ευρώ το μήνα, αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορείτε να φανταστείτε πρέπει να πληρώνουν όλες τους τις δαπάνες, τα εξοδά τους, να πληρώνουν για τη διατροφή τους, τα φάρμακα. Και πραγματικά τους καταλυστεύουν από αυτό που έχτισαν οι ίδιοι μέσα από τα προγράμματα ιδιωτικοποίησης στην ε, Βουλγαρία υπό την αιγίδα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου. Πρέπει, είναι τραγικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μα όταν μιλάμε για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στου άλλους εγγεγραμμένου αγορητέ, ξεκινώντα από τον κύριο Μαν που έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012 το έκανε Ευρωπαϊκό Έτος Συμμετοχής των Ηλικιωμένων στην Ενεργό Ζωή και ε, ανταποκρίθηκε στην πρόταση της Επιτροπής μας. Είναι σημαντικό. Πρόταση που έρχεται τη σωστή στιγμή. Υπάρχουν άνθρωποι άνω των 80 που και αυξάνει το αριθμό τους που είναι υγιείς. Από το 2010 μέχρι το 2030 θα υπάρξει αύξηση αυτού του ποσοστού κατά 60%. Στην ερώτηση της Επιτροπής ε, ζητούμε ναι, την Κομισιόν να μας μιλήσει για τα υπέρ και τα κατά της φροντίδας όπως παρουσιάζεται σήμερα και να προβεί στη συναγωγή συμπερασμάτων. Όλο και περισσότερες οικογένειες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη φροντίδα. Δεν υπάρχουν ε, τα απαραίτητα πρόσωπα. Όμως ε, καλό είναι το ε, προσωπικό, το ειδικευμένο να μπορεί γρήγορα να αντικαθίσταται ε, πολλές φορές ε, ένας είναι ο υπεύθυνο για τη φροντίδα. Τώρα για τη δικαιοσύνη απέναντι στις γενναίες κάλεσα τα κράτη-μέλη να ε, θεσπίσουν καλύτερα συστήματα ελέγχου γιατί όσοι χρειάζονται φροντίδα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι και η αξιοπρέπειά τους θα παραμείνει αλόβητη. Ε, καλό είναι να υπάρχουν ελάχιστες ε, παροχές για τη μακροπρόθεσμη φροντίδα ανεξάρτητα από την ηλικία, την, την κατάσταση της υγείας, ε, τον κίνδυνο για την υγεία. Θα πρέπει όλοι να έχουν καλή φροντίδα γιατί δεν είναι βάρος ηλικιωμένοι. Η εμπειρία τους, ε, τα επιτεύγματά τους διαμόρφωσαν την κοινωνία μας. Δεν μπορεί να επιτρέπεται να τους αφήσουμε μόνους με τα προβλήματά τους. Να αξιοποιήσουμε το χρονικό διάστημα μέχρι το 2012 για να δημιουργήσουμε πολλές προϋποθέσεις, ώστε η πολιτική, τα μέσα και η κοινή γνώμη να ασχοληθούν με, την, ε, ε, με τους ηλικιωμένους στην εργοζωή. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όλων μας υπέρ μιας βιώσιμης ε, φροντίδας η οποία δεν θα προσανατολίζεται μόνο προς το κόστος. Κύριε Ράπτη, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Α, θέλω να πω το εξής. Όταν μιλάμε όλοι μας σε αυτή την αίθουσα για τους ηλικιωμένου, ίσως να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι κάποια στιγμή μπορεί και εμείς οι ίδιοι να γίνουμε ηλικιωμένοι. Να φτάσουμε στα 80, στα 90 και στα 100 χρόνια έχουμε φανταστεί ποτέ πώς θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται. οι άνθρωποι αυτοί που έχουν κάποια ηλικία είναι οι άνθρωποι που μας έδωσαν ζωή είναι οι άνθρωποι που μας έδωσαν πολιτισμό είναι οι άνθρωποι που είναι η προσωπική μας περιουσία εντός εισαγωγικών. η μακροπρόθεσμη φροντίδα των ηλικιωμένων έχει την ηθική διάσταση την κοινωνική διάσταση αλλά έχει και την οικονομική διάσταση διότι κάθε υπερήλικας που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα σημαίνει ότι μειώνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων μελών της οικογένειάς του ενώ παράλληλα εάν θεσπίσουμε ένα πρόγραμμα φροντίδας μπορεί και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. αυτά όλα ας τα σκεφτούμε κυρία επίτροπε και ας δώσουμε μια κατεύθυνση στα κράτη μέλη. ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους μεταφραστές που μας δίνουν την ευκαιρία να εκφράζουμε την άποψή μας μετά τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Τσικάου έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σύμφωνα με πρόσφατες στατιστικές, μέχρι το 2050 ο αριθμός των ατόμων πέραν των 65 θα αυξηθεί κατά 70% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 170% θα είναι το ποσοστό των ατόμων που θα έχει ξεπεράσει τα 80. Άρα θα έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά. Θα πρέπει να ευρεθούν λύσεις ε, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ε, ε, ανάγκες φροντίδας όλων αυτών των συστήματων, να το προβλέψει στα συστήματα κοινοτική προστασίας και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Θα πρέπει να ευρεθούν επίση λύσει για να υπάρχουν και οι απαραίτητε ρυθμίσει σε θέματα στέγασης και σε θέματα μεταφορών. Θα ήθελα να χαιρετήσω την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τα δικαιώματα των ε, επιβατών για τα άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς και για τους ηλικιωμένους που μετακινούνται με οποιαδήποτε μέσο μεταφοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την προσέγγιση της προσοχής. Δίνω το λόγο στον κύριο Νικολάζικ. Πρόεδρε. Ε, το θέμα είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις δημογραφικές αλλαγές που πιέζουν και τους προϋπολογισμούς. Καλό είναι μεταξύ άλλων να έχουμε βιώσιμες πολιτικές ενώ αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, κατάργηση των διακρίσεων Θεωρώ σημαντικό το θέμα της αλληλεγγύης. Εδώ θα πρέπει οι φροντίζοντες του ε, τους ηλικιωμένους να ε, έχουν και κάποια επιδόματα, κάποια οικονομική υποστήριξη. Καλό είναι λοιπόν εδώ να γίνει μια ανταλλαγή καταξιωμένων πρακτικών σε αυτό το τομέα. Ως γιατρός θέλω να πω ότι ε, είμαι κατά των εντολών μη ανάνυψης, γιατί αυτό αντιφάσκει προς τα ανθρώπινα δικαιω... θεμελιώδη δικαιώματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζαμπόσκα έχει το λόγο για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Autori položili Európskej komisii 10 otázok. Medzigeneračnej... Ευχαριστώ πολύ. Η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών ε, είναι σημαντική. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα όμως σε αυτό το περίπλοκο θέμα. Προηγουμένως ε, συζητούσαμε για την επιρροή της Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Γιατί δεν προτείνει η Κομισιόν τα κράτη-μέλη να ε, Δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ε, φροντίδα στην οικογένεια. Γιατί ένα, κράτος, ένα μέλος της οικογένειας ε, δεν μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα και να υποστηρίζεται οικονομικά. με δεδομένο ότι δεν μπορεί και να εργάζεται και ταυτόχρονα να αναλάβει μια τέτοια φροντίδα γιατί θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις εφόσον μιλάμε για το πνεύμα της αλληλεγγύης. Θα ήταν πολύ περισσότερο οι άνθρωποι αν γινόντουσαν ίδια τα πράγματα. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον τελευταίο αγορητή, τον κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το ότι συζητάμε αυτό το θέμα είναι κάτι πολύ επίκαιρο. Είναι μεγάλο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Και ευχαριστώ την κυρία Λίν που υπογράμμισε ιδιαίτερα τα προβλήματα που υφίσταται σε αυτή την όπως αποκαλείται πολιτισμένη κοινωνία όσον αφορά την κακομεταχείριση των ηλικιωμένων. Επίσης ο Επίτροπος έδωσε μια πλήρη περιγραφή, περιέγραψε τους στόχους, τις προκλήσεις και τις λύσεις. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό σαν μια δυνατότητα. Δυνατότητα να επιτρέψουμε στον κόσμο να ξεπεράσουν τα όρια της ηλικία που έχουν τεθεί τώρα και να μπορούν να ταξιδεύουν και να συμβάλλουν επίσης και στον τουρισμό έχουμε την πρόκληση να, φροντίσουν, ε, να φροντίζονται αυτοί οι άνθρωποι στο σπίτι του επί μακρόν και βεβαίω και ε, φροντίδα στα ιδρύματα που παρέχεται. Δεν έχουν ληφθεί υπόψη οικονομική συνεισφορά εκείνων που προσέχουν του ηλικιωμένου και θα πρέπει να κάνουμε κάτι ούτω ώστε να υπάρχει ε, σωστή περίθαρψη των ηλικιωμένων στα επόμενα χρόνια. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ο Επίτροπος, ο κύριος Άντορ, έχει το λόγο. Έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, να επαναλάβω αυτά που είπαμε στην αρχή της συζήτηση για την ε, ποικιμορφία της Ευρώπης. Έχουμε 27 κράτη-μέλη με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες, ε, υλικές υποδομές και συνθήκες και γι' αυτό κυρίως ε, εργάζεται στα στο πλαίσιο ε, της ε, ισότητας με αυστηρότερη νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση και θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα αυτό μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το οποίο πρόσφατα συζητήσαμε πανηλημμένα το θέμα. Ένα κέριο ζήτημα ε, που αφορά και τη συναγωγή συμπερασμάτων πώς ε, η φροντίδα, η μακροπρόθεσμη συνδέεται με την ατζέντα μας, πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εδώ. Αλλά έχουμε και το καθήκον να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στην ατζέντα των ε, δεξιοτήτων, προσόντων και να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για την εκπαίδευση, κατάρτιση, την ε, δημιουργία μεγαλύτερου αποθέματος ατόμων που μπορούν να αναλάβουν τη φροντίδα με επαγγελματισμό. Είναι ανοιχτό το ερώτημα σε ποιο βαθμό πρέπει να ρυθμίσουμε τις υπηρεσίες αυτές, γιατί όπως ελέγχθη, μεγάλο κομμάτι της φροντίδας που παρέχεται είναι άτυπη γίνεται από συγγενείς μέσα στην οικογένεια. Η ρύθμιση λοιπόν, ε, η δημιουργία προτύπων, η δημιουργία προϋποθέσεων μέσα στο πλαίσιο των οικογενειών και των συγγενών είναι ε, πολύ προβληματικό θέμα γιατί ενώ ρυθμίζουμε αυτό, αυτές τις εργασίες θα αυξάναμε τις δαπάνες, θα προέκυπταν θέματα φορολογίας και θα αντιμετωπίζαμε πολλά διέξοδα. Δεν υπάρχει εύκολη απάντηση, ενώ υπάρχει πιεστική ανάγκη βελτίωσης των συνθήκων εκείνων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και που είναι εξαρτημένη από τη μακροπρόθεσμη φροντίδα. Παράλληλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ορισμένα πράγματα σε αυτούς που τους φροντίζουν. Πρέπει να συλλέξουμε και να διαβάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές, χρησιμοποιώντας και την ανοιχτή μέθοδο του συντονισμού επίσης. Μπορώ να πω αυτή την περασμένη ώρα ότι σε λίγες ώρες θα συναντήσω ορισμένους υπουργούς από τη βελγική κυβέρνηση στη Λιέγη, στην διάσκεψη για τις συντάξεις, και αυτή θα είναι μια καλή ευκαιρία για να μεταφέρω τους λόγους του Κοινοβουλίου επί του θέματος αυτού και να το συνδέσω με το έργο μας ε, για τις συντάξεις, γιατί είναι αλληλένδετα τα θέματα αυτά και οι ανησυχίες που αφορούν ένα επαρκές εισόδημα ε, και κοινωνική ασφάλιση επαρκή για τους ηλικιωμένους. Έχουμε και πιο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα να δώσουμε συνέχεια στο έργο μας με τις συντάξεις, με μια ε, σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του δημογραφικού. Η Ουγγαρία και η Πολωνία, οι επόμενες προεδρίες, εξίσου ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Και τώρα διερευνούμε το κατάλληλο πλαίσιο για τα παραδοτέα, όπως λέμε, και μετά θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Έτος Συμμετοχής των Ηλικιωμένων στην Ενεργό Δεν είναι μόνο για την απασχόληση αυτό, ούτε είναι μόνο θέμα παράτασης η συνταξιδοτικής κάλυψης. αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε την υγεία, να διατηρήσουμε την ικανότητα διαβίου, μάθησης και παροχής εκπαίδευσης από τα διάφορα ιδρύματα για να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής. Αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε και θα συνεχίσουμε το έργο μας. Ε, είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις, αλλά με την ηθική δέσμευση που είναι κοινή για όλους μας, νομίζω ότι θα ε, έχουμε αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Δίνω το λόγο στη συντάκτρια την κυρία Λίν ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που πήραν το λόγο και να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο για αυτά που μας είπε απόψε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά αυτό που απέρεσα από τη συζήτηση επίσης είναι η έκκληση που έβαλα στο προφορικό ερώτημα και στην, για το διδολογικό κώδικα που ο Τόμας Μάν ανέφεραν και άλλοι. Δεν μιλάμε εδώ για νομοθεσία όπως προανέφερα και νομίζω το καλό παράδειγμα της Βουλγαρίας για κάποιον που ζητάμε 100 ευρώ το μήνα και πρέπει να πληρώσει για μακροπρόθεσμη περίθαλψη ήταν ένα από του λόγου για του οποίου χρειαζόμαστε αυτό το λειτουργικό κώδικα. Ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να πληρούν κάποιε ελάχιστε προδιαγραφέ. Και το ίδιο ε, για τι εντολέ να μην γίνεται για την επαναφορά στη ζωή ε, όταν κάποιο περνά μια καρδιακή κρίση. Λοιπόν, και πρέπει να γίνεται αλλαγή βελτίστων πρακτικών και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει πολλή δουλειά για να μας βοηθήσει να μπορέσουμε να δώσουμε τις βέλτιστες, ε, να δώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών μελών και ευχαριστώ και τους διερμηνείς που ξεπέρασαν την, το όριο της 12ης νυχτερινής. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Σας λέω ότι έλαβα πρόταση ψηφίσματος προ το τέλο τη συζητήσεω, πέρα τη συζητήσεω. Ψηφοφορία θα λάβει χώρα την 5η στι 12. Σα ευχαριστώ και ευχαριστώ και εγώ του διερμηνεί. Επόμενη συνεδρίαση αύριο Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου από τις 9 μέχρι 13 και από τις 15 μέχρι τις 18 και από τις 21 μέχρι τις 24.